Καλώ Καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Στην Επιτροπή αυτή θέτουμε τους καταναλωτές στο ίδιο επίπεδο, τουλάχιστον στο ίδιο, αν όχι σε ανώτερο, με τους παρόχους υπηρεσιών. Επομένως, με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε την Επίτροπο Βέρα Γιουροβά, Κατά την, άποψή μας, οι αρμοδιότητες της για τη δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα φύλων είναι πολύ σημαντικές. Εμείς θα βάλουμε μπροστά μας τους καταναλωτές. Ευχαριστούμε που ήρθατε να μας συναντήσετε. Ο σκοπός της συνάντησης είναι να συζητήσουμε την πρόοδο του, που έχει γίνει στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν και στις πρωτοβουλίες να ανταλλάξουμε απόψεις για τους εκρεμείς νομοθετικούς φακέλους και να δούμε τις προτεραιότητες για τη χρονιά που μας περιμένει. Θα κάνει μια εισαγωγική δήλωση επίτροπος. Εξήγησα ότι διάφοροι ευρωβουλευτές είναι μακριά εκτός ε, κοινοβουλίου σε διάφορες ε, αποστολές, αντιπροσωπείες κτλ. αλλά σχεδόν ε, οι πέντε μεγαλύτερες εθνικές αντιπροσωπείες είναι πολύ καλά εκπροσωπημένες. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ την Επιτροπή ΙΜΚΟ για τη συνεργασία και για την πρόσκληση που μου επίφθηνε για να μιλήσω σε αυτόν τον διαρθρωμένο διάλογο. Αν θυμάστε την ακρόασή μου, και σε άλλες συνεδριάσεις που είχα έρθει στην ΕΝΚΟ είχα υποσχεθεί ότι θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Όχι μόνο μέσω τέτοιων συνεδριάσεων, αλλά και στο διάμεσο διάστημα με συμβουλευτικέ συναντήσεις, συμβουλευτικού χαρακτήρα δηλαδή συναντήσεις, θα είμαστε πάντα σε επαφή. Κάθε ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσουμε και να ακούσω τις απόψει σα, τη χρησιμοποιώ. Σε όλη την θητεία μου θα ακούω τη φωνή των καταναλωτών, αλλά και των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων και ευπαθών καταναλωτών. Θέλω να έχουν περισσότερες επιλογές, περισσότερη προστασία και περισσότερη εμπιστοσύνη. Η λιδία λήθος, όποτε παίρνουμε νέες πρωτοβουλίες, είναι η εμπιστοσύνη. Επομένως θα πρέπει σε όλες τις προσπάθειές μας να έχουμε μπροστάριδες στους καταναλωτές. Τους τελευταίους μήνες ε, σημειώσαμε πρόοδο σε διάφορες πρωτοβουλίες που θα δώσουν απτά ωφέλη στους καταναλωτές. Να σας τονίσω η πρόταση για την Ενεργειακή Ένωση που παρουσίασε η Κομισιόν στις 25 Φεβρουαρίου, όπου βάζουμε τους καταναλωτές στο κέντρο. Θέλουμε καταναλωτές να ασχολούνται με την ενέργεια και με θέματα μετάβασης προς νέες τεχνολογίες για να μειώσουν ε, τους λογαριασμούς τους, να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά και να είμαστε σίγουροι ότι προστατεύονται οι ευπαθείς καταναλωτές. Μαζί με, τον... με τη Σεσίλια Μάλστρομ, τη συνάδελφό μου, θα εξασφαλίσω τα συμφέροντα των καταναλωτών στις διαπραγματεύσεις για το TTIP με τις ΗΠΑ. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε μία συμφωνία η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών και τι ανησυχίε του. Οι, οι συμφωνίε συμφωνίε θα πρέπει να μειώσουν τι τιμέ και να δώσουν ποιοτικέ θέσει απασχόληση. Αυτό ακριβώ θα πρέπει να μα εξασφαλίσει το TTIP και να προστατεύσει παράλληλα τα συμφέροντα των καταναλωτών. Ένα άλλο στοιχείο είναι να δώσουμε ε, εξουσία στους καταναλωτές στην ε, ψηφιακή ενιαία αγορά που είναι προτεραιότητα για αυτή την Κομισιόν. Θα ε, δρομολογήσουμε σε λίγες εβδομάδες στρατηγική για αυτό το θέμα. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις προσανατολισμού ανατολισμού ε, στο Σώμα των Επιτρόπων. Εγώ θα συνεισφέρω σε υπό διάφορε έννοιε αυτή τη στρατηγική. Από συμβάσει, προστασία των δεδομένων, ε, εργαλεία ε, σύγκριση μέχρι θέματα υπολογιστικού νέφους. Θέλω να απλουστεύσουμε τους κανόνες των, για τους καταναλωτές για αγορές στο διαδίκτυο. Η ψηφιακή ενιαία αγορά έχει την, το δυναμικό να γίνει η ατμομηχανή για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2014, το 15% των αγορών των καταναλωτών ε, έκανε τα ψώνια τους καταναλωτές μάλλον ε, από άλλες χώρες. Ενώ 44% το έκαναν εσωτερικά και μόνο το 5% των επιχειρήσεων ε, πούλησαν τα προϊόντα τους διασυνοριακά online θα πρέπει ακόμα να αναπτύξουμε το δυναμικό και να το εκμεταλλευτούμε αυτό το δυναμικό της ενιαίας αγοράς. Έχουμε δηλαδή πολλές δυνατότητες ανεκμετάλλευτες. Οι σημερινοί κανόνες για τις άδικους συμβατικούς όρους δεν προστατεύουν επαρκώς καταναλωτές για το προβληματικό περιεχόμενο των συμβάσεων αυτών ε, που αφορούν αγορές στο διαδίκτυο. Ε, επίσης για ελαττωματικά προϊόντα δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν αρχίσει να φτιάχνουν τέτοιου κανόνε για τα ψηφιακά προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καλύψει αυτό το νομικό κενό πριν έχουμε 28 διαφορετικούς κανόνες από τα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε την δυνατότητα τώρα να υποβάλουμε τον κανονισμό για το ψηφιακό περιεχόμενο. Είμαι ανοιχτή σε διαφορετικές ε, επιλογές. Θέλουμε να έχουμε δίκαιες λύσεις που θα δώσουν καταναλωτές πρόσβαση στην ψηφιακή ενιαία αγορά χωρίς ε, να βαράνουμε υπερβολικά τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις και τη δικαιοσύνη, για τις μικρομεσαίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συχνά είναι θύματα σε παραπλανητικές ε, πρακτικές διαφήμισης, ειδικά online και ειδικά όταν μιλάμε για συναλλαγές στο διαδίκτυο. Η οδηγία του 2006 για την παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση δεν είναι αποτελεσματική και δεν είναι εναργή σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή διάσταση. Γι' αυτό παρουσιάσαμε μια αναθεώρηση πέρυσι που δυστυχώς καθυστερήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών εκλογών. Καθυστέρησε, συγγνώμη, λόγω των ευρωπαϊκών εκλογών. Θέλουμε να ανισχύσουμε την νομική ασφάλεια και να εξασφαλίσουμε καλύτερη προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εναντίον απατών ε, στο μάρκετινγκ, στη διαφήμιση κτλ. Και θέλουμε να απαγορεύσουμε διάφορες παραπλανητικές πρακτικές. Σε δεύτερη φάση θέλουμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή διασυνοριακά. Η πολιτική για τους καταναλωτές δεν αφορά μόνο τα νομοθετικά θέματα, αλλά και τα πρακτικά εργαλεία, ε, την επίλυση των διαφορών. Πριν από δύο εβδομάδες, οι συνάδελφοί μου παρουσίασαν στο Κοινοβούλιο ένα μοντέλο της, ε, της πλατφόρμας για την επιγραμμική επίλυση διαφορών. Με χαρά έμαθα ότι αυτή η δοκιμή πήγε πολύ καλά. Έλαβα πληροφορίες ότι υπήρχαν 20 συμμετέχοντες και αν υπάρχει ενδιαφέρον μπορούμε να κάνουμε ακόμα μια προσπάθεια για να δουν κι άλλοι. Τον Ιανουάριο του 2016 θα είναι λειτουργική η πλατφόρμα και θα φέρει μεγάλες αλλαγές στη σχέση μεταξύ των Ευρωπαίων καταναλωτών και των εμπόρων ε, επιγραμμικά. Η πλατφόρμα αυτή επίλυση ε, διαφορών online θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών καθώ και την αξιοπιστία των εμπόρων. Η ίδια η αρχή των εξχρονισμένων κανόνων αφορά την πρότασή μα για την, το πακέτο για του ταξιδιώτε. Ε, δουλεύουμε μαζί με τους συνομοθέτες για να φτάσουμε στην τελική συμφωνία. Είμαι ευγνώμων για τη δουλειά σας και θέλω να ευχαριστήσω κυρίω τον την εισηγήτρια την κυρία Λάγκεν, τους σκιώδεις εισηγητές και βεβαίως ε, την πρόεδρο την κυρία Φόρντ, καθώς και τη Λετωνική Προεδρία. Βασίζομαι στην ε, αδιάλειπτη ε, υποστήριξή σας, στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, τόσο ώστε να έχουμε συμφωνία τους επόμενους μήνες. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της θητείας μου θα ήθελα να δώσω μεγάλη έμφαση στο πώς η νομοθεσία για τους καταναλωτές εφαρμόζεται στην πράξη. Η προστασία, η συνεργασία των κρατών μελών για θέματα προστασίας των καταναλωτών είναι βασικό στοιχείο και χρειαζόμαστε να την εφαρμόσουμε και στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Ετοιμάζοντας την ανθεώρηση του κανονισμού για την συνεργασία με σκοπό την προστασία των καταναλωτών, μελετούμε τι καλύτερε λύσει για να ενισχύσουμε τι δυνατότητε των κρατών μελών για να σταματήσουν τι επιγραμμικέ παραβάσει και να αντιμετωπίσουν πιο γρήγορα τι εκτεταμένε αυτέ παραβάσει στο διαδίκτυο. Κύριε Ευρωβουλευτέ, γνωρίζω τον επόμενο μήνα είναι η επέτειο τη πρώτη νομοθεσία για του καταναλωτέ πριν από 40 χρόνια. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 1975, του Απριλίου 1975, για ένα πρόγραμμα για την προστασία των καταναλωτών και μια ενημερωτική πολιτική, μίλησε για πέντε βασικά δικαιώματα για πρώτη φορά. Το δικαίωμα στην προστασία, τη υγείας και τη ασφάλειας, το δικαίωμα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, το δικαίωμα ένδικων μέσων, το δικαίωμα στην πληροφόρηση και στην εκπαίδευση και το δικαίωμα στην εκπροσώπηση. Συν το χρόνο και βαθμία σημειώσαμε πρόοδο προς αυτά τα βασικά δικαιώματα και στη συνθήκη και σε μεμονωμένα νομοθετήματα που αποτελούν σήμερα το κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών. Τα 400 γενέθλια της νομοθεσίας αυτής είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να σκεφτούμε πού θέλουμε να εστιάσουμε στο μέλλον. Θα ήθελα να έχουμε μια προσέγγιση στραμμένη προς το μέλλον για την προστασία των καταναλωτών, κατάλληλη για τον 21ο αιώνα. Και η υποστήριξή σας είναι ζωτική σημασία. Θέλω να συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά μαζί σας για τα επόμενα κεφάλαια αυτής της ιστορίας. Και εξίσου σημαντικό θέλω να συνεχίσω την επικοινωνία ε, για τα επιτεύγματά μου. Επιτεύγματα μας έχουμε πολλές ευκαιρίες ε, φέτος, όπως το, τη Σύνοδο ε, για τους καταναλωτές τον Ιούνιο, για να συζητήσουμε την πολιτική για τους καταναλωτές του μέλλοντος. Και έχετε και την ευκαιρία να συζητήσετε αυτά τα θέματα σήμερα μαζί μου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much for covering... Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που καλύψατε όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές. Ή αυτούς τους, ε, τους αντικαθαστούν και μετά να ακούσουμε τις υπόλοιπες ομάδες. Ποιος ε, εκπροσωπεί την κυρία Γκέπχαρτ. Η κυρία Τον νομίζω αντικαθιστάτε τον Ανδρέα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Επιτροπή, που βρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μας και που μας παρουσιάσατε τη δουλειά σας, το έργο σας έως τώρα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό το χαρτοφυλάκιό σας και στην ε, Επιτροπή μας είμαστε πραγματικά πολύ ικανοποιημένοι με τις επιτυχίες σας. Ήθελα καταρχάς να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι οι σχέσεις των καταναλωτών θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες στη ψηφιακή αγορά. Μιλάμε για μία αγορά ψηφιακή Εμεί εμείς ε, προσπαθούμε να κάνουμε τους πάντες να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε αυτά. Το ίδιο ισχύει και για τους ε, καταναλωτές. Είτε μιλάμε για την ψηφιακή αγορά, είτε για την πραγματική αγορά, θα πρέπει να έχουν την ίδια προστασία. θα έχουμε και την 40η επέτειο της πρώτης νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. 40 χρόνια. Θα πρέπει κάπως να το γιορτάσουμε μαζί. Είπατε ότι θα ενημερώσουμε τον κόσμο, θα πληροφορήσουμε για τις επιτυχίες μας. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα μεγάλο μειονέκτημα, ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Φυσικά έχουμε πετύχει πολλά πράγματα, αλλά το γνωρίζουν οι καταναλωτές. Η πολιτική επικοινωνία των θεσμικών οργάνων πραγματικά έχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και ελπίζω ειλικρινά εσείς να το πετύχετε αυτό. Να καταφέρετε να ενημερώσετε τον κόσμο πέρα από τις Βρυξέλλες, προκειμένου να ξέρει τι δικαιώματα έχει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις επιχειρήσεις, για την οικονομία. Άμα δεν γνωρίζουν οι καταναλωτές τι δικαιώματα έχουν, δεν εμπιστεύονται τις επιχειρήσεις και έτσι δεν ωφελούνται και οι επιχειρήσεις ίδιες. Δεν έχουν το κέρδος που θα μπορούσαν να έχουν. Χρειάζονται λοιπόν οι καταναλωτές επιχειρήσεις που λειτουργούν σωστά και στις οποίες να μπορούν να υπολογίζουν. Τώρα, για την επίλυση διαφορών ε, σε διαφορά τις ε, επιγραμμικές της online αγορές. Είχαμε μια καλή ιδέα και θεωρώ ότι ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και καταδεικνύει συγκεκριμένες λύσεις για τους καταναλωτές. Αυτό θα ενισχύσει την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ένα πράγμα που θα πρέπει να βελτιώσουμε και το έχω παρακολουθήσει πολύ στενά είναι το εξής. Το θέμα της γλώσσας. Ένα τμήμα της μετάφρασης λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, αλλά ένα άλλο τμήμα ειλικρινά δεν τα πήγε καθόλου καλά. Όταν συζητήσαμε με τους καταναλωτές και μας λένε στις διάφορες χώρες τι διακριτική μεταχείριση δέχονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν αντιμετωπίζεται συνήθω από την Επιτροπή από την πλευρά του καταναλωτή, επειδή κάποια προϊόντα δέχονται αρνητική μεταχείριση. Το ίδιο ισχύει και για τι μηχανέ αναζήτηση στο διαδίκτυο από πλευρά καταναλωτή. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις που παραμένουν για την πρόσβαση στα προϊόντα αυτά. και η έλλειψη ενό κοινού δικαίου για τι αγοραπολισίες. Τεράστιο πρόβλημα. Προκειμένου να μπορέσει ο καταναλωτή να επωφελείται σωστά από την ψηφιακή αγορά. Και όχι μόνο σε ψηφιακό επίπεδο, αλλά και στις ε, πραγματικέ, στις φυσικές, τις συνδεσμένες παραδοσιακές αγοραπολισίες, αλλά και ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον. Αλλά για παράδειγμα εγώ δεν μπορώ να δω στη χώρα μου το House of Cards, τη σειρά που μου αγαπώ, που τη βλέπω μόνο στο Βέλγιο. Ε, κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμη Επιτροπέ. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να σας καλωσορίσω εδώ στην Επιτροπή μας και να σας μιλήσω στην πιτρική μας γλώσσα να σας ευχαριστήσω για τα εισαγωγικά σας λόγια και σας ευχαριστώ για την, την τριπλή προτεραιότητα που αναφέρατε σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές, την ανάγκη να έχουν εμπιστοσύνη, να έχουν νομική βεβαιότητα και το καθεξής. Θα ήθελα να περιοριστώ ωστόσο σε δύο ερωτήσεις. Ένα ζήτημα το έθεσε και η προηγούμενη ομιλητρία, η κυρία Τούν. Τη διακριτική μεταχείριση των καταναλωτών ανάλογα με τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο προέλευσής τους. Αυτή η διακριτική μεταχείριση πώς μπορεί να αποφευχθεί προκειμένου να προσεγγίσουν και οι προσωπικές μας εμπειρίες Δεν είναι περιθωριακό αυτό το φαινόμενο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κεντρική καταγραφή των υπηρεσιών και των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ποιότητες των προϊόντων που πολλούνται στις διάφορες χώρες. Εσείς μιλήσατε για την εμπιστοσύνη. Ρωτώ, συμφωνείτε ότι η διακριτική μεταχείριση κάποιων καταναλωτών πλήττει την εμπιστοσύνη τους στα προϊόντα και τι σκοπεύετε να κάνετε. Ποια είναι η ατζέντα σας σε σχέση και με το έργο των συναδέλφων σας. Ένα δεύτερο ερώτημα τώρα. σε ό,τι αφορά ενεχόμενη καταγγελία από πλευρά του καταναλωτή μιας παράνομης δραστηριότητα. Όπω ξέρετε υπάρχει μια οριζόντια νομοθεσία για την συλλογική σύμβαση, τις συλλογικές αγωγές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 δημοσίευσε μια σύσταση και μίλησε για εθελούσιες αγωγές. Πόσα θέλω να ξέρω έχουν εφαρμόσει αυτό το μηχανισμό για τη συλλογική νομική προστασία και τα συστήματα αυτά είναι συμβατά το ένα με το άλλο στην ιστορική αγορά. Αν ο μηχανισμός αυτός δεν έχει πετύχει τον στόχο του, θα μπορούσατε να φανταστείτε μια νέα νομοθετική πρόταση και όλα αυτά θα με ενδιαφέραν και σε σχέση με το ενδεχόμενο ευρωπαϊκό δίκαιο για τις αγοραπολισίες. Simple. Πολύ απλά έχετε το λόγο. Ίσως να περάσουμε σε όλες τις πολιτικές ομάδες στον πρώτο γύρο για τους συντηρητικούς, Ντόλτον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Καταρχάς με ικανοποίηση σας άκουσα να μιλάτε για την ωφέλεια που μπορεί να έχει το TTIP για τους ε, καταναλωτές, γιατί φοβάμαι ότι στα πλαίσια της γενικότερης συζήτησης για άλλα θέματα του TTIP ε, δεν ακούγονται πολλά ιδιαίτερα καλά για τους ε, καταναλωτές. Κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την ασφάλεια, τον κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Υποτίθεται ότι έχετε κάνει μία ανάλυση για το άρθρο 7 για την υποχρεωτική αναγραφή του κράτους προέλευσης. Δεν ξέρω πώς πηγαίνει η μελέτη αυτή την οποία κάνατε. Και σχετικά με την ενιαία ψηφιακή αγορά. Πράγματι οι νέοι κανονισμοί δημιουργούν προβλήματα στις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις να πολλούν τα προϊόντα τους. Και φοβάμαι ότι προσπαθώντας να λύσουμε τα προβλήματα που υπονομεύουν την ψηφιακή αγορά σε ορισμένους τομείς δημιουργούμε νέα σε άλλους τομείς. Θα επαναλάβω λίγο αυτά τα οποία είπαν και οι συντονιστές από τις άλλες ομάδες τώρα πλέον. Έχουμε ένα θέμα. Όταν κάποιος αγοράζει ένα ψηφιακό αγαθό, δεν συνειδητοποιούν το προϊόν ότι δεν μπορούν να το μεταφέρουν και να το χρησιμοποιήσουν όταν πηγαίνουν σε μια άλλη ε, περιοχή. Ε, σαν παράδειγμα είπε ε, η κυρία Χόχενστάιν το παράδειγμα του House of Cards. Για μένα είναι το cricket στην τηλεόραση ε, και είναι υποχρεωτικό ουσιαστικά. Αν δεν μπορείς νόμιμα να βλέπεις στην τηλεόραση κάτι, προσπαθείς να βρεις με πειρατικό τρόπο θα έλεγα την εκπομπή της επιθυμίας σου. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει θα πρέπει να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει στον κόσμο να πάρει το περιεχόμενο το οποίο επιθυμεί και να ρυθμίσουμε ανάλογα και τις άδειε, οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν. Λοιπόν, πρέπει να κατανοήσουν τους περιορισμούς της αδειοδοτήσης ε, των εκπομπών από οι καταναλωτές. Στα πλαίσια λοιπόν του διαλόγου για τις άδειε ε, για το περιεχόμενο το τηλεοπτικό, το ψηφιακό, ε, μπορείτε να ενημερώσετε περισσότερο για το ποιες είναι οι περιοριστικές διατάξεις στον τομέα της κυκλοφορίας αυτών αυτού του περιεχομένου του ψηφιακού. Από τη φιλελεύθερη ομάδα η κυρία Τσαράνσοβα. Ευχαριστώ την ε, Επίτροπο, πράγματι έθεσε πάρα πολλά θέματα και αυτό το κατανοήσατε ήδη και από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των προηγούμενων συναδέλφων. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, το ένα αφορά το TTIP και το άλλο αφορά την ενιαία ψηφιακή αγορά. Για το TTIP είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα το πρωί. Προσπαθούμε να επεξεργαστούμε μια έκθεση για το TTIP και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπατε για τη σημασία που έχει αυτή η συμφωνία για τους καταναλωτές μας. Το μήνυμα ακριβώς της Επιτροπής αυτής, αυτή την κατεύθυνση θα ακολουθεί. Στα πλαίσια της ενιαίας ψηφιακής αγοράς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πρόκληση και σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι και εσείς σαν υπεύθυνοι για την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να ακούγεται η φωνή σας ε, στα πλαίσια του καθορισμού της στρατηγικής για την ψηφιακή αγορά. Μία ερώτηση που συνδέεται με τα θέματα αυτά είναι η λεγόμενη ε, διαμοιρασμένη οικονομική δραστηριότητα. Πολλοί χρησιμοποιούν σήμερα το eBay σαν παράδειγμα ε, για να κλείσουν επίσης τις διακοπές τους Υπάρχει μια ψηφιακή οικονομία λοιπόν η οποία αναπτύσσεται και εν πολύ αντικαθιστά κάποια παραδοσιακά μοντέλα της αγοράς. Μπορείτε να μας δώσετε λοιπόν κάποια παραδείγματα για την προστασία των καταναλωτών που συμμετέχουν στα νέα αυτά πρότυπα. Ένας ακόμα και μετά θα μιλήσετε εσείς κυρία Τζούροβα. Ευχαριστώ Βίκη. Ευχαριστώ και την Επίτροπο που είναι παρούσα σήμερα εδώ. Και την ευχαριστώ επίσης και για μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση. Έχω τέσσερις ερωτήσεις για τα θέματα στα οποία ήδη αναφερθήκατε. Το ένα είναι η ενέργεια. Θα πρέπει να πω ότι σαν καταναλωτής, όταν πηγαίνω να αγοράσω, μου αρέσει να πηγαίνω να αγοράσω ένα σακάκι, αλλά είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο το να προσπαθήσω να κάνω επιλογή μέσα από τις διαφημίσεις ε, ε, επιχειρήσεων ε, παραγωγής και προσφοράς ενέργειας. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κατανοήσει κανείς τα επιχειρήματα. Υπάρχουν βέβαια κάποια site συγκριτικά, τα οποία όμως δεν είναι ουδέτερα και γι' αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο για ένα καταναλωτή να μπορέσει να πάρει μια ισορροπημένη απόφαση για το ποιε είναι οι επιχειρήσεις από τις οποίες θα πρέπει σε εισαγωγικά να ψωνίσει. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να απλοποιήσει τα πράγματα για τον καταναλωτή για να ισχύσει έτσι και τις ικανότητες του καταναλωτή να απλοποιήσει α, τις επιλογές του. Τώρα για το TTIP. Είστε υπεύθυνο και για τα θέματα της δικαιοσύνης και γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, ασχολείται με το θέμα της οικονομίας της ευρωπαϊκής νομικής τάξης. Αυτό είχε τεθεί και στα πλαίσια της ε, πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τι σημαίνει αυτό για το TTIP. Αν πάρετε την απόφαση σαν παράδειγμα για του δικαστηρίου, την απόφαση του δικαστηρίου για την οδηγία ε, για τους καταναλωτές. Θα δείτε ότι αλλάζει τους κανόνες για το μέλλον και επηρεάζει ίσως αρνητικά τελικά τις ε, επενδύσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να ισχύσει και για το IDS και το θέμα εδώ είναι ότι η απονομή δικαιοσύνης ε, θα παρεμποδιστεί από την απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και από ό,τι γνωρίζω έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται. Λοιπόν, ποια θα είναι η σχέση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την αυτονομία ε, της Ευρωπαϊκής Νομικής Τάξης και τις ρυθμίσεις για τις, ε, για διευθετήσεις που ισχύουν στα πλαίσια του TTIP. Ένα άλλο θέμα. Στη Γαλλία, σαν παράδειγμα, μπορεί να αποκτήσει κανείς μια διεύθυνση .fr εφόσον έχει την έδρα της επιχείρησής του στη Γαλλία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν σαν καταναλωτής ε, ψάξεις μια επιχείρηση στην Γαλλία, πολλές φορές δεν θα βρεις τη διεύθυνση αυτή γιατί είναι ε, πολύ συνηθισμένο να σου προσφέρονται τα αποτελέσματα άλλου τύπου επιχειρήσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα διαδεδομένων. Και για την παραπλανητική διαφήμιση επίσης είναι εξαιρετικό το ότι θέλετε να ασχοληθείτε και με αυτό το θέμα. Μας έχετε υποσχεθεί ότι θα αναλάβετε δράση και χαίρομαι που θα το κάνετε. Μία σύσταση από πλευράς μου. Νομίζω ότι οι κανόνες είναι ένα πράγμα. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο για τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν κάποιους κανόνες. Στην Ολλανδία σαν παράδειγμα Έχουμε ε, ε, μια υπηρεσία η οποία βοηθά τις επιχειρήσεις να καταγγέλουν τις απάτες και να προστατεύονται από αυτές. αν υπήρχε ένα δίκτυο αυτών των υπηρεσιών, τότε θα μπορούσαμε να συλλέξουμε πάρα πολλές ε, πληροφορίες για το ποιες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τις παραπλανητικές αυτές πρακτικές. Λοιπόν, θα μπορούσαμε λίγο ε, να δούμε τι γίνεται και με το θέμα της επιβολής των προτάσεων τις οποίες κάνετε, όχι μόνο το περιεχόμενό τους. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε να απαντήσει η, Κομισ... η Επίτροπος ε, όλες τις ερωτήσεις. Όταν ο καθένας μας υποβάλλει πέντε ερωτήσεις, θα προσπαθήσει πάντως να απαντήσει κάποιες από αυτές. Ε, και νομίζω ότι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει και ως καλές ιδέες. Σας ευχαριστώ. Μια και μπορώ να μιλήσω τσέχικα, θα μιλήσω τσέχικα, που είναι και η μετρική μου γλώσσα. Έτσι θα είμαι και πιο συγκεκριμένη, πιο λακωνική. Σας ευχαριστώ όλους για τις ιδέες σας. Με εμπνέουν. Δεν, δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις ως πολιτικός ε, υποτίθεται ότι μπορώ να λέω αυτά που θέλω να λέω. Οι πολιτικοί αποφεύγουν κάποιες ερωτήσεις, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να ακολουθήσω εδώ το, τη σειρά. Ε, για αυτό που είπε η κυρία Τούν, για την ιδέα της καλύτερης επικοινωνίας. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου θέματα, η επικοινωνία. Και ο κόσμος στο ιδιωτικό μου γραφείο το ξέρει πάρα πολύ καλά πόση σημασία δίνω σε αυτό. Θέλουμε οι καταναλωτέ να είναι ενημέροι, θέλουμε να αποφασίζουμε τα λόγου γνώσεως, θέλουμε όλοι να ξέρουν τι κάνουμε εμείς επίσης και τι ετοιμάζουμε. Μπορώ να σας δώσω πολύ επικαιροποιημένα παραδείγματα. Κάτι που συνέβη σήμερα μάλιστα. Μπορώ να σας αναφέρω. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για τις 31 λεγόμενες αθέμητες πρακτικές, έτσι τις λέμε. Αθέμητες, 31 είναι αυτές οι αθέμητες πρακτικές και κάνουμε μία εκστρατεία ενημέρωσης. Μας απασχολούν ιδιαιτέρως οι ευπαθείς και ηλικιωμένοι πολίτες και γενικά οι πολίτες οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουν κατά ανάγκη τους κινδύνους ε, που ενέχουν ορισμένες συναλλαγές. Είναι καθήκον μας να τους ενημερώσουμε. Ένα άλλο παράδειγμα. Κάτι άλλο το οποίο θα, με το οποίο θα παρενοχλήσω τους συναδέλφους μου, γιατί με απασχολεί πολύ και θα το προωθήσω. Τον Ιανουάριο θα ξεκινήσουμε το σύστημα ε, επιγραμμικής επίλυσης διαφορών, όπως ξέρετε, τον Ιανουάριο του 2016 δηλαδή. Θα είναι ένας τρόπος για να μπορεί ο κόσμος να επιλύει τα προβλήματά του. Αν έχει λάβει, ας πούμε, ε, κάποιο αγαθό, το οποίο δεν λειτουργεί, δεν δουλεύει. Αυτή η πλατφόρμα που λέγεται ODR θα είναι η κατάλληλη πλατφόρμα για να επιληθούν οι διαφορές. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μάθει ο κόσμος την 1η Ιανουαρίου. Καλό θα ήταν να το ξέρει ήδη εκ των προτέρων και ειδικά όταν κάνει τις χριστουγεννιάτικες αγορές του του 2015 δηλαδή. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την εκστρατεία ενημέρωσης νωρίς, τον Οκτώβριο, Νοέμβριο κτλ. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τότε οι καταναλωτές ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το σύστημα επίλυσης διαφορών από 1η Ιανουαρίου του 2016. Φυσικά ξέρουμε ότι θα υπάρξουν κάποια προβληματάκια, αλλά τουλάχιστον θα υπάρχει αυτό το σύστημα. Δεύτερο, το επόμενο θέμα. Μεταφράσεις και γλώσσες σε αυτό το σύστημα επίλυσης διαφορών αυτή την πλατφόρμα που λέγεται ODR. Θα υπάρχει ένα σύστημα αυτόματης μετάφρασης. Θα υπάρχουν πάντως προβλήματα, γιατί ε, το μηχάνημα δεν ξέρει πώς να μεταφράζει πάντα από μία γλώσσα σε οποιαδήποτε. Υπάρχουν κάποια ζεύγη γλωσσών ε, που είναι λίγο πιο προβληματικά. Όμως ασχολούμαστε αυτό το θέμα και θα ασχοληθούμε περαιτέρω και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις μεταφράσεις. Μπορεί επίσης να καλέσουμε και κάποιου μεταφραστέ, να κάνουν οι ίδιοι ε, τις μεταφράσεις όταν υπάρχει κανένα άλλο τρόπο. Επομένω, η τελική μετάφραση, η τελική ας πούμε, η καλύτερη, πιο αυθεντική, θα, την κάνει, θα γίνει από άνθρωπο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια προβληματάκια με την πλατφόρμα αυτή την ODR. Προσπαθούμε να βρούμε πρακτικέ και ρεαλιστικέ λύσει, ούτω ώστε όλε οι γλώσσε να καλύπτονται. Μην ανησυχείτε λοιπόν. Ε, αυτή η εκστρατεία ενημέρωση θα υπάρξει. Μίλησα για την πλατφόρμα ODR. Το επόμενο σημείο. Για να δω ποιο θα είναι. Αν θα έχουμε μεγαλύτερες ε, και περισσότερες επιλογές οι καταναλωτές. Το House of Cards. Αυτό το project. Α, αυτό έχει να κάνει με το θέμα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Και το θέμα της ε, νέας ε, νομοθεσίας που καλύπτει την αγορά ψηφιακού περιεχομένου. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, θέλουμε να έχουμε κοινέ νομοθεσίες στα κράτη-μέλη. Έχουμε τρία κράτη-μέλη που έχουν νομοθεσία και όλα τα υπόλοιπα κενό. Θέλουμε να προωθήσουμε την αρμόνιση σε αυτό το τομέα. Ο κύριος Ντάλτον θέλει να εξασφαλίσει ότι όταν οι καταναλωτές αγοράζουν ψηφιακό περιεχόμενο, να ξέρουν τι αγοράζουν. Να ξέρουν τα όρια. Αν είναι άδεια, ας πούμε, και τα λοιπά να ξέρουμε ποια είναι τα όρια. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι περιορισμοί και πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όταν πληρώνουν οι καταναλωτές ε, ξέρουν τι θα πάρουν για αυτό που πληρώνουν. Έχω πάει σε διάφορες ε, συνεδριάσεις, σε διάφορες συζητήσεις και μία από τις πιο σεξι συζητήσεις για τις οποίες μιλούσε η Ντίτα Χαρανζόβα αφορούσε ακριβώς την ενιαία ψηφιακή αγορά. Και κυρίως το θέμα των αγορών ψηφιακού περιεχομένου online. Εμείς έχουμε πολύ ξεκάθαρες ιδέες. Έχουμε σχετική νομοθεσία που την προωθούμε. Έχουμε επίσης και υλικά αγαθά. Ασχολούμαστε και με αυτά στην Επιτροπή. Μαζί με την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και συνεργαζόμαστε με τον Αντιπρόεδρο Άντρου Σάντσιπ, που έχει την ε, γενικότερη ευθύνη και εποπτεία για, την για το ψηφιακό θεματολόγιο. Κάνουμε συζητήσεις λοιπόν με τους συναδέλφους αυτούς για τα δικαιώματα των καταναλωτών, τις επιλογές των καταναλωτών στο ίντερνετ. Ήταν απόφευκτο να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή ε, το, δίκαιο για, το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο για τις ε, αγορές αποσύρθηκε. Αυτή τη στιγμή αποσύρθηκε, έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε με το θέμα της ασφάλειας δικαίου. Έπρεπε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία, ούτω ώστε ο καταναλωτής να αγοράζει στο ίντερνετ να έχει εμπιστοσύνη σε αυτό που αγοράζει. Επίσης μας ανησυχούσε και το θέμα του άχθους που βαραίνει τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να το μειώσουμε ή δυνατόν. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν την κατάλληλη ισορροπία. Θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Η κυρία Μπιενκόφσκα υπέβαλε κάποιες προτάσεις. Μιλάει για τη χρήση του δικαίου που διέπει τις ε, λειτουργίες του εμπόρου. Αλλά κοιτάξτε, Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν κάποιες, κάποια δέσμη κανόνων που δεν μπορεί να αγνοηθεί, την οποία θα εμπιστεύεται ο καταναλωτής. Γιατί όλα θα τα κάνουμε για τους καταναλωτές που δεν είναι δικηγόροι, έτσι, που δεν διαβάζουν κατά ανάγκη τα ψηλά των συμβάσεων που υπογράφουν. Ορισμένοι δεν διαβάζουν καν τη σύμβαση που, που, αγοράζουν, ε, που χρησιμοποιούν θέλουν οι περισσότεροι όταν αγοράσουν κάτι στο ίντερνετ να το πάρουν αυτό το οποίο φαντάζονται ότι αγοράζουν και δεν θα υπάρξουν άσχημες εκπλήξεις. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές ας πούμε σε αυτό που αγοράζει στο ίντερνετ ο καταναλωτής ε, στην Τσεχία, στη Δανία, στην Τσεχία κτλ. Θα πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών παντού. Το έχω πει κατ' επανάληψη. Δεν θέλουμε να υποσκάψουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και δεν θέλουμε να μειώσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών στο ίντερνετ. Ούτε θέλω να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δικαιώματα των καταναλωτών στο ίντερνετ και εκτός ίντερνετ. Θέλω να υπάρχουν υψηλά πρότυπα, είτε αγοράζει κανείς στο ίντερνετ, είτε εκτός στον πραγματικό κόσμο. Έχουμε αυτή την νομοθεσία για τις πωλήσει online και παίζουμε με την ιδέα ενός μοντέλου συμβάσεων που θα σέβεται όλους αυτούς τους κανόνες για τους οποίους σας μίλησα προηγουμένως. Κοιτάμε τις συμβάσεις που αυτή τη στιγμή διέπουν τις ε, επιγραμμικές ε, συναλλαγές στην Ευρώπη και ανακαλύψαμε το 60% των συναλλαγών online από τους Ευρωπαίους καταναλωτές διέπονται αυτή τη στιγμή από το καλιφορνέζικο δίκαιο. Το 60%. Εδώ στην Ευρώπη δηλαδή αγοράζουμε online με βάση μια νομοθεσία που υπάρχει κάπου στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές είναι οι συμβάσεις των καταναλωτών ε, online με βάση οποίες αγοράζουν τις περισσότερες φορές καταναλωτές, εδώ, στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να ξικιώνται αρκετά με όλα αυτά. Και θα πρέπει, πιστεύω, να ξαναδούμε λιγάκι αυτούς τους κανόνες. Καθώς προσπαθούμε να εισαγάγουμε ευρωπαϊκούς κανόνες, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι στο ύψος των θεμητών προσδοκιών των Ευρωπαίων καταναλωτών. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μια συζήτηση στο Σώμα των Επιτρόπων με αυτές τις ιδέες. Εγώ θα μιλήσω για την προστασία των καταναλωτών ε, όταν αυτοί αγοράζουν στο διαδίκτυο. Θα πω τις ιδέες μου και σε έξι μήνες θα υποβάλουμε μία νέα πρόταση νομοθετήματος καθώς και μία μελέτη αντικτύπου. Επομένως σέβομαι το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε ήδη τεθεί ας πούμε. Τώρα πάμε στο TTIP. Έγινε μια ερώτηση την κυρία Σενάλοβα. Για μια προσπάθεια αποτίμησης των ένδικων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Των ομαδικών ένδικων μέσων. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. 23 κράτη-μέλη έχουν εισάγει στην νομοθεσία τους κάποια μορφή τέτοιων ένδικων μέσων. Δεν θα τα διαβάσω από τα κρατη είναι η μεγάλη πλειοψηφία, 23 από τα 28 κρατη Θέλουμε μέχρι τον Ιούλιο του 2017 να αξιολογήσουμε αυτά τα νομικά συστήματα των 23 αυτών κρατών μελών. Και αν οι συστάσεις μας δεν ήταν επαρκείς και τα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, ανταποκριθεί με επαρκή τρόπο, τότε θα προτείνουμε νέα νομοθεσία. Δεν ξέρω αν θα είναι οδηγία ή καονισμός τώρα, θα το αποφασίσουμε αργότερα. Επόμενο σημείο. Τιτ-τυπ. Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση με την κυρία Μάλστρομ στο Σώμα των Επιτρόπων το Φεβρουάριο. Εγώ προσεγγίζω το θέμα του TTIP όχι μόνο από τη σκοπιά της προστασίας των δεδομένων, αλλά και την προστασία των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά την επίλυση των προβλημάτων των επενδυτών, υπάρχουν τέσσερις κανόνες που έχουμε συμφωνήσει. Το δικαίωμα ρυθμίσεων τη δημιουργία και λειτουργία ενός δικαστηρίου διατησίας, τη σχέση μεταξύ ε, των εθνικών εγχώριων δικαστικών συστημάτων και του συστήματος επίλυσης διαφορών επενδυτών κρατών και η αναθεώρηση του συστήματος ISDS και ο μηχανισμός ε, προσφυγών. Τέσσερις κανόνες λοιπόν συνολικά και εξακολουθεί να ισχύει ότι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα είναι εκείνα τα οποία θα συνεχίσουν να εκδικάζουν τις υποθέσεις αυτές. Δεν θα γίνεται όλα μέσω διατησίας. Για τις ε, άδειες, το TTIP, συμφωνία TTIP. η κοινή οικονομία. Μεγάλη είναι η πρόκληση αυτή για μας. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ρύθμιση. Αφενός λοιπόν ε, υπάρχει μια έκκληση για μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή. Αλλά στο σενάριο αυτό Ποιο είναι ο καταναλωτή που χρειάζεται προστασία, γιατί οι, προστασία, οι καταναλωτές που ξεκινούν τη διαδικασία αυτή ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν ότι δεν υπάρχει κάποια ρυθμιστική προστασία. Νομίζω λοιπόν ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται ότι αν χρησιμοποιούν την φορολογική υπηρεσία αυτή, ή αν ανταλλάσσουν τα σπίτια τους, πολύ απλά θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι υπεύθυνοι για αυτό που κάνουν. Ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που ενέχονται. Πρόκειται για νέες μορφές καταναλωτικής συμπεριφοράς και όλα αυτά αποτελούν απόρρια της ψηφιακής ε, επανάστασης. Ο τρόπος συμπεριφοράς των καταναλωτών, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αξιολογούμε σε ό,τι αφορά και το τι θα γίνει στο μέλλον. Και θα ήθελα να κάνω εδώ πέρα μία μικρή παρένθεση, αν θέλετε. Όταν ο κόσμος ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα, οι κοινωνιολόγοι ήταν πολύ ανήσυχοι και έλεγαν ότι πρόκειται για έναν τρόπο να εκτονώνει την ενέργειά του η πλειονότητα. Η πλειονότητα η οποία ω τότε ήταν σιωπηλή απέκτησε φωνή. Και αυτό λοιπόν σημαίνει σήμερα και με την οικονομία. Ο κόσμος παίρνει την οικονομία στα χέρια του. Χρησιμοποιεί τι ψηφιακέ. Ε, συνδέσεις για να ανταλλάξει σπίτια, να ανταλλάξει διαμερίσματα για τις δέσκοπές του. Και θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες ε, είναι οι τάσεις που διακρίνονται, τι κάνει ο κόσμος. Αν αποφασίσουμε δε να νομοθετήσουμε, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η νομοθεσία δεν πρόκειται να καταπνίξει αυτόν τον αυτορμητισμό στη συμπεριφορά του κόσμου. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε τον κόσμο να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρέμβουμε και να παρεμποδίσουμε αυτή την ψηφιακή οικονομία. Αυτή είναι η ψηφιακή οικονομία και φυσικά υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Και όποιος ε, έχει μια επιχείρηση online θα πρέπει να σέβεται τους κανόνες αυτούς. Αλλά πριν αρχίσουμε να νομοθετούμε, ας κοιτάξουμε τι νομοθετούμε ακριβώς, ποια είναι η κατάσταση που μας οδηγεί και τι θα πρέπει να γίνει. Γιατί όλα αυτά είναι καινούργια, όπως είπα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κατάλογος των ομιλητών περιλαμβάνει τους εξής. Then Ildiko Galpelch, then um, Christophe Chaldemosa, then Lucy Anderson, then Virginie Rosary. Is there anybody? Okay. Anybody else? Κανείς άλλος? Όχι. Ωραία. Η Άννα Μαρία λοιπόν έχει το λόγο. Εν συντομία όμως, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. καλύψετε πάρα πολλά στην ε, παρουσίασή σας και θα θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας, για την ελεύθερη επιλογή των καταναλωτών, για την ψηφιακή αγορά, την οποία, στην οποία προσβλέπουμε όλοι στην ε, ανακοίνωση. Όπως ξέρετε, το ηλεκτρονικό εμπόριο τα πηγαίνει πολύ καλύτερα στα σύνορα της κάθε χώρας. Τα προβλήματα είναι πολύ πιο μεγάλα μεταξύ των χωρών μιλήσατε για, την, ε, για τον εξυγχρονισμό της προστασίας του καταναλωτή. Τι λέτε όμως, θα ξαναξεκινήσετε να κάνετε αναθεώρηση της οδηγίας για την προστασία των καταναλωτών. Για τις διάφορες συμβάσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο, γιατί αυτό θα προκαλούσε πρόβλημα στην ουδετερότητα του δικτύου. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια απλούστευση. Δεν νομίζω ότι αυτό θα ωφελούσε τον καταναλωτή αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε. Είπατε ότι θα εστιαστείτε στην πλήρη εφαρμογή της ε, συνθήκης, της ε, νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της πραγματικής διαφήμισης και χαίρομαι, χαίρομαι που θέλετε να το ξαναθέσετε επιτάπητος. Και αυτό περιλαμβάνει ένα τμήμα της προστασίας του καταναλωτή. Προτίθεστε να ασχοληθείτε με το θέμα της επιθετικής ε, διαφήμισης κατά των παιδιών ως ευάλωτοι καταναλωτές. καταναλωτές. Ε, για το θέμα της περιαγωγής. Ξέρετε ότι το Συμβούλιο έχει τοποθετηθεί διαφορετικά από το Κοινοβούλιο για το πότε θα πρέπει να καταργηθεί ή κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν ανώτατα όρια για το roaming, για την περιεγωγή. Το κόστος που θα σημαίνει αυτό για τις υποδομές και κάποιοι ανησυχούν ότι θα αυξηθούν οι τιμές ε, για τους ε, καταναλωτές. Με ποιο χρονοδιάγραμμα θα κινηθείτε. Μιλήσατε για τον κανονισμό και την προστασία των δεδομένων. Και πάλι έχουμε πρόβλημα με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Ποιο είναι λοιπόν το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων. Ελπίζω να περάσει αυτό που είπατε, μια καλύτερη ισορροπία, αλλά και καλύτερη πρόσβαση προς πελαστημότητα για τις μικρές επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας πιο πολύ υπόψη το γεγονός ότι θα πρέπει να αντέξει στο μέλλον αυτή η διαμόρφωση. Τελευταίο ζήτημα, δεν αναφερθήκατε στην ισότητα μεταξύ των φύλων που περιλαμβάνεται το χαρτοφυλόκια σας. Ξέρω ότι υπάρχουν προγράμματα προώθησης των γυναικών και της επιχειρηματικότητας των ε, γυναικών, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόσβαση των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα στην ψηφιακή αγορά. Ευχαριστώ και τελείωσα. Η Πρόεδρος. Οι γυναίκες στη δική μας επιτροπή στην παρούσα φάση ξεπερνούν τους άντρες. 9 γυναίκες, 5 άντρες. Και αυτό επειδή συμμετέχουμε πιο πολύ παρά το γεγονός ότι οι άνδρες οι οποίοι παρίστανται είναι πάρα πολύ δραστήριοι. Πρέπει να είμαι, καταλαβαίνετε, ευγενής και προς τις δύο πλευρές. Η κυρία Γκάλ Πέλτς. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ ε, την Επίτροπο τα θέματα με τα οποία ασχολούνται, ασχολείται έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχουν πάρα πολλοί παροχείς, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές, υπάρχουν όμως και κάποια μειονεκτήματα, υπάρχουν νομικά προβλήματα, θέματα προστασίας του καταναλωτή κτλ. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους θα θέλατε να συγκεντρώσετε την προσοχή σας στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών στο πλαίσιο της ψηφιακής αγοράς. Είπατε ότι έχετε ήδη προχωρήσει σε κάποια βήματα. Ποια είναι. Θα συνεργαστείτε επίσης με τον κύριο Έτιγκερ για τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να είναι φιλικές προς τους καταναλωτές. Πιστεύετε ότι μπορείτε να ξεκινήσετε μια αυτόνομη νομοθετική διαδικασία για την προστασία των καταναλωτών. Είχα και επιπλέον ερωτήσεις μετά από αυτά που είπε και η Αν Μαρή. Συνεπώς κάποιες από αυτές θα σας τις θέσω. Τα άρθρα για την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να κυκλοφορήσουν ε, και να ενημερώνουν σωστά τους καταναλωτές. Έχετε ε, αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα βοηθήσουν τον καταναλωτή να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη και μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα και ίσως και μια ρυθμιστική αρχή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Σχέλντελ Μόσερ. Ευχαριστώ. Επίτροπε, πάντα εσείς θέλετε να είσαστε σε διάλογο με την Επιτροπή μας και με το σύνολο του Κοινοβουλίου. Ένα θέμα που δεν μας απασχόλησε σήμερα είναι η ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω γιατί βρίσκεστε στην αρχή της εντολής σας. Μιλήσατε όμως για την ψηφιακή ατζέντα. Και θα ήθελα να μου πείτε αν μία από τις λύσεις τις οποίες προτείνεται στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων, το λεγόμενο made in δηλαδή, ε, μπορεί να επιληθεί μέσω ε, ψηφιακών τρόπων. Δηλαδή είναι κάτι στο οποίο μπορείτε να σκεφτείτε να υπάρξει μια σφραγίδα στο προϊόν ψηφιακή. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να μειώσει και το κόστος των επιχειρήσεων. Να μπορεί κανείς ε, να κάνει ένα σκάν ε, πάνω σε ένα πακέτο, σε ένα προϊόν έτσι ώστε να βλέπει κανείς τι, ε, σε τι τομείς προστατεύεται με την αγορά του προϊόντος. Αναφερθήκατε στο TTIP. Το θέμα εδώ συνδέεται βέβαια με την εμπορική συμφωνία για τη χώρα προέλευσης. Υπάρχει και η συμφωνία ΣΕΤΑ η οποία θα επηρεάσει το TIP. Έχετε αναλύσει τις πιθανές συνέπειες ε, αυτής της ε, σύνδεσης. Lucy Anderson. Thank you. Anderson. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Άκουσα αυτά τα οποία μας είπατε για την προσφυγή στη δικαιοσύνη και για τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί. Είναι όμως επίσης σαφές ότι θεωρητικά τουλάχιστον η πρόσβαση στην δικαιοσύνη ε, γίνεται αντικείμενο εγγύησης του άρθρου 47 αλλά είναι και κάτι το οποίο συνδέεται με το δίκαιο των καταναλωτών. Προσπαθήσαμε να δούμε σε επίπεδο διαδικασίας αν τα δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται σύμφωνα με τις αποφάσεις και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τι βήματα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, είναι σαφές ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε μπορέσει να βρούμε μία λύση και αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Μία αναθεώρηση λοιπόν συνολική σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων είναι κάτι το προαπαιτούμενο έτσι ώστε να προοδεύσουμε. Και τι γίνεται με το στοχολόγιο το οποίο είχατε διαμορφώσει στον τομέα της δικαιοσύνης. Είχατε στείλει τα ερωτηματολόγια, αλλά δεν πήραμε απαντήσεις. Ε, αναρωτιέμαι λοιπόν αν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Και τέλος για την εκστρατεία Keep Me Posted. Δεν είναι μόνο μια ψηφιακή εκστρατεία, αλλά καλεί τους καταναλωτές να επιλέγουν ε, εάν επιθυμούν να δέχονται ε, κάποιες πληροφορίες για τα προϊόντα τους, όχι μόνο ψηφιακά, αλλά και ε, σε χαρτί. Ευχαριστώ Πρόεδρε λέει η κυρία Ροζιέρ. Ευχαριστώ και την Επίτροπο για την παρουσία της. Πολλά ερωτηματικά υπάρχουν γύρω από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να θέσω α, κάποιες ερωτήσεις. Η περίμετρος, αν θέλετε, των προτάσεών σας περιορίζεται στην προστασία των καταναλωτών ή και σε ευρύτερα θέματα. Ε, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να νομιμοποιήσει μια διαφοροποιημένη προστασία του καταναλωτή και ποια είναι η φύση της πρότασης. Θα είναι ένα νέο 21ο καθεστώς, μια μέγιστη εναρμόνιση, μια ελάχιστη εναρμόνιση με εθνικά καθεστώτα διαφοροποιούμενα μεταξύ τους. Και σε αυτή την περίπτωση ποια είναι η βασική αρχή η οποία θα εφαρμόζεται. Ε, θα είναι η έδρα του πολιτή, η έδρα του καταναλωτή. Ε, υπάρχουν πολλές απορίες. Τώρα για τα πολιτιστικά προϊόντα, όπως γνωρίζετε η πρόσβαση στα πολιτιστικά προϊόντα απασχολεί το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας λοιπόν στο ότι σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα γίνονται κάποιες συζητήσεις οι οποίες δεν ανήκουν εκεί η συζήτηση για πρόσβαση ε, σε ψηφιακό προϊόν διασυνοριακά. Είναι κάτι το οποίο ε, δεν έχει άμεση σχέση μόνο με το δικαίωμα το πνευματικό του δημιουργού, αλλά κυρίως με την άδεια εκπομπής ψηφιακού περιεχομένου του συγκεκριμένης επιχείρησης. Σε ορισμένους τομείς υπάρχουν πανευρωπαϊκές άδειε, αλλά η αγορά σήμερα είναι διαμορφωμένη σε επίπεδο ε, εθνικό και δεν έχουν συμφέρον οι μεγάλοι διανομής περιεχομένου ψηφιακού να αλλάξει το υπάρχον καθεστώς. Όταν κάποιος όμως αποκτήσει ε, τα δικαιώματα σε μία χώρα μπορεί να πρέπει μάλλον να έχει τη δυνατότητα να ασκεί ε, τα δικαιώματα αυτά που έχει αγοράσει και σε άλλες χώρες. Βλέπουμε τι γίνεται με το ψηφιακό περιεχόμενο του, του Αμερικανικού διαδικτύου. Ξέρουμε επίσης ότι ε, αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ευεργετικά για την ε, συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα για την παραγωγή στις Ηνωμένε Πολιτείες και αυτό έχει άμεση σχέση βέβαια και με τις αμοιβέ των καλλιτεχνών. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ επίρροπε, Ο κ. Ριμούντ. Κατά την απάντηση στον πρώτο γύρο είπατε ότι θα προσπαθήσατε να απαντήσετε πάρα πολύ ξεκάθαρα στις ερωτήσεις και θα προσπαθήσετε να τις αποφύγετε. Μία λοιπόν μικρή ερώτηση έχω να κάνω, την οποία και έχω θέσει και σε άλλες υπηρεσίες, αλλά ποτέ δεν έχω πάρει ουσιαστικά μία απάντηση. Στο θέμα λοιπόν του κατά πόσον ε, είναι σημαντική για σας η προστασία του καταναλωτή, φυσικά θα απαντήσετε ναι. Και το κατά πόσον ε, θέλετε αυτό να το προστατεύσετε στο TTIP, σίγουρα θα μας απαντήσετε καταφατικά και κατά πόσον θα πρέπει να προστατεύσουμε στις διαπραγματεύσεις των καταναλωτή στην Ευρώπη, φυσικά θα μας απαντήσετε καταφατικά. Αυτό που διαπιστώνουμε ωστόσο είναι ότι στο ΣΕΤΑ στις περιγραφές προέλευσης 1.400 ε, υπάρχουν ε, στην Ευρώπη προστατεύονται μόνο 150 επωνυμίες προέλευσης, μόνο 145 μάλλον από τις 1400. Πώς το εξηγείτε λοιπόν αυτό, πώς το εξηγείτε αυτό στον Ευρωπαίο καταναλωτή που θέλετε να τον προστατεύσετε και κατά τρίτον, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα συμβεί το ίδιο στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας TTIP. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Ακούσατε την άποψη των μελών της Επιτροπής ότι είμαστε εδώ για να φροντίσουμε ότι θα ακουστεί η φωνή των καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη και σε όλο το Κοινοβούλιο και ότι ελπίζουμε να καταστήσουμε λειτουργική την ενιαία αγορά προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτέ να μπορέσουν να ευμερίσουν και στα 28 κράτη-μέλη. Είναι άρα πολύ σημαντικό για μα να ακουστεί η φωνή του καταναλωτή. Να μην ξεχνάμε ποια είναι η φωνή του καταναλωτή και να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτέ δεν θα έχουν λιγότερη προστασία στην ενιαία αγορά από αυτή που έχουν συνηθίσει στι εγχώριε αγορέ του ή στην ψηφιακή αγορά σε σχέση με την παραδοσιακή αγορά. Πρώτη ερώτηση λοιπόν, όταν θα, θα, θα μας βοηθήσετε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι διαφορετική η αντιμετώπιση της προστασίας του καταναλωτή στον ψηφιακό από τον πραγματικό κόσμο και ότι μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες ότι όταν υπογράφουμε συμφωνίες η προστασία του δεν θα διακυβευτεί λόγω των συμφωνιών αυτών. Κατά δεύτερον, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οργανώσεις σας θα βάλουν πάνω από όλα τη φωνή του καταναλωτή. Μπορείτε λοιπόν να διασφαλίσετε ότι στην εσωτερική αναδιάταξη και αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνεχίσετε να ακούγεται η φωνή του καταναλωτή. Θα σας υποστηρίξουμε κι εμείς, άρα θα μας υποστηρίξετε κι εσείς για να εισακούετε η φωνή του καταναλωτή. Ακόμα και σε άλλες επιτροπές θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχνάμε τον καταναλωτή. Για τα συγκεκριμένα ζητήματα τώρα για τα δικαιώματα του καταναλωτή και για τον ψηφιακό κόσμο. Καταλαβαίνουμε ότι σε κάποια περιβάλλοντα δεν υπάρχει προστασία καταναλωτή. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το Κοινοβούλιο όμως θα εκτιμήσει τις προτάσεις αυτές. Αλλά ούτε οι ενώσεις του καταναλωτή δεν πίστευαν ότι υπάρχει επαρκής προστασία από πλευράς τους. Θα μας πάρει πολλά χρόνια όμως να υπάρξει πήρε μάλλον πολλά χρόνια η διαπραγμάτευση τη σχετική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή. Τι προτείνετε? Αρχικά τουλάχιστον να υπάρξει ενό είδου σύμβαση για να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και παράλληλα να εξετάσουμε κατά πόσο χρειάζεται νομοθετική λύση. Τα μοντέλα συμβάσεων θεωρώ ότι θα βοηθούσαν άμεσα για το θέμα του TTIP. Μιλήσαμε το θέμα, για το θέμα του ISDS, της επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους. Μπορείτε να φέσετε όμως το θέμα του TTIP, τη διαφάνεια πάνω απ' όλα, για να μην υπάρχει διαιτησία του επενδυτή. Γιατί υπάρχει η φημολογία ότι η διαιτησία γίνεται πάντα και κλεισμένων των θυρών. Δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό, θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια. Και μία ίσως πονηρή ερώτηση. Η Επιτροπή μας πάντα θέλει καλύτερη νομοθεσία και καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και θέλουμε ένα τμήμα της Επιτροπής μας να εστιαστεί σε θέματα εφαρμογής. Θα θέλατε να μας ξαναεπισκεφτείτε με μέλη της υπηρεσίας σας για να δούμε πως κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα ο online μηχανισμός επίλυσης διαφορών, πώς ε, μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα και αυτό και άλλα συστήματα και όχι απαραίτητα εσείς αυτοπροσώπους, αλλά ίσως θα μπορούσατε να αποστείλετε τους επιλογνώμονές σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητήσουμε τέτοια θέματα, για παράδειγμα της ε, επίλυσης διαφορών. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας, θα καθυστερήσουμε λίγο. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από το τέλος και από την ερώτηση της κυρίας Φόρντ. Η πολιτική των καταναλωτών όπως τη βλέπουμε εμείς είναι θέμα εμπιστοσύνη. Είναι και θέμα θεμητών προσδοκιών. Ό,τι και να κάνουμε θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ε, θα πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το θέμα δεν είναι να νομοθετούμε για να νομοθετούμε. Έχουμε πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς μεγάλη νομοθετική παραγωγή. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με τη νέα νομοθετική ε, ρύθμιση. Πριν περάσουμε όμως τη νέα νομοθετική ρύθμιση, θα πρέπει να βεβαιωθούμε για την συμπεριφορά του καταναλωτή και τις λύσεις τις οποίες έχουν καταλήξει οι υπόλοιποι τομείς. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται στη συμπεριφορά των ιδίων των αγορών. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω να προωθήσω νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες βασίζονται στην ε, ορθή πρακτική και δεν παρεμποδίζουν την ανάπτυξη ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα. Σχετικά τώρα με το mainstreaming και την προστασία των καταναλωτών σε όλους τους τομείς. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει στο γραφείο μου και στη Γενική Διεύθυνση είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι με το λεγόμενο mainstreaming. Λέγουν λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει καμία νομοθετική ρύθμιση η οποία δεν θα λαμβάνει υπόψη αυτά τα οποία ισχύουν για την προστασία του καταναλωτή. Δηλαδή θα αξιολογούμε και θα εκτιμούμε πάντα θέματα όπως η ενέργεια του Επιτρόπου κ. Σεύκοβιτς, είναι ένας καλός τομέας στον οποίο παρενέβημε ακριβώς λόγω της εμπιστοσύνης την οποία θα πρέπει να τρέφει ο καταναλωτής προς τις ρυθμίσεις μας. Η οδηγία τώρα για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Όπως γνωρίζετε θα υπάρξει μια αναθεώρηση η οποία είναι συνέπεια της εξέτασης του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Τίθεται και το θέμα του εναρμονισμού των ρυθμίσεων για τις διαδικτυακές πωλήσει. Είναι μία οδός και αυτή. Έχουμε κάποιους βασικούς κανόνες ενισχύ, έχουμε κάποιες βασικές αρχές για τις υποχρεώσεις τις λεγόμενες προσυμβατικές, και για τις υποχρεώσεις οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ισχύω της σύμβασης. Αλλά εκεί όπου έχουμε πολλά προβλήματα είναι ε, σε σχέση με την αποκατάσταση των ζημιών που μπορεί να προκληθούν από μια σύμβαση. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε κάποιες νεότερες προτάσεις στα πλαίσια της νέας ψηφιακής αγοράς. Αυτό είναι μια πρώτη λύση και θα προχωρήσουμε σε αυτό ε, στα πλαίσια της αναθεώρησης. Το θέμα είναι να καλύψουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν. Αγαπητά μέλη λοιπόν, εγώ θέλω να ακολουθήσω τις προτάσεις σας, αλλά με προειδοποίησαν κάποιοι συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και η Κοράτσα Μπίλτ, για το μακρόχρονο των διαδικασιών αυτών. Θα απαιτηθεί πάρα πολύς χρόνος, ώσπου να ε, υπάρξει μια τελική διευθέτηση. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος για μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση από το μακρόχρονο της διαδικασίας. Αν ακολουθήσουμε το δρόμο του ρεφίτ, εάν πράγματι λοιπόν επιλέξουμε την οδό της αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, τότε μπορούμε να βρούμε μια λύση σε εθελοντική βάση. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα ονομάζαμε μια σύγχρονη συμβατική διαδικασία. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα συζητήσουμε, θα προτείνουμε ένα πρότυπο συμβόλαιο ε, στους ε, εμπόρους, στους επιχειρηματίες ε, της ψηφιακής αγοράς και θα υποδείξουμε λοιπόν και στον καταναλωτή ότι στα πλαίσια της σύμβασης την οποία προβαίνει υπάρχει μία κάποια εγγύηση νομική, υπάρχει μία κάποια πιστοποίηση για τον συγκεκριμένο έμπορο. Υπάρχουν δηλαδή ορισμένοι κανόνες οι οποίοι θα γίνουν σεβαστοί. Αυτή δεν είναι μια νομοθετική λύση βέβαια. Είναι μια λύση η οποία θα απαιτήσει πάρα πολύ προσπάθεια στον τομέα της ενημέρωσης, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε εφόσον ε, μακρόχρονη όπως είπα είναι η διαδικασία και μας καθυστερήσει. Λοιπόν αυτό είναι το σχέδιο που έχουμε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σκοπεύουμε εμείς να ξεπεράσουμε την δυσκολία της νομοθετικής διαδικασίας. Πρέπει κάτι να κάνουμε και νομίζω ότι οι εμπορευόμενοι στην ψηφιακή αγορά θα καταλάβουν ότι θα τους βοηθήσουμε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών όχι σε μία χώρα μόνο αλλά και στις 28. Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Γνωρίζω ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Λοιπόν, για την ισότητα των φύλων τα είπαμε, για τον αθέμητο ανταγωνισμό, για τους ευάλωτους καταναλωτές, ιδιαίτερα τα παιδιά, όλα αυτά μας απασχολούν. Βλέπουμε εμείς τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας τα οποία χρειάζονται οι διαφορετικές κατηγορίες των καταναλωτών. Έχουμε μια μελέτη, περιμένουμε να ετοιμαστεί τον Απρίλιο και ανάλογα θα προχωρήσουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε, να βοηθήσουμε να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των προβλημάτων και για την παραπλανητική διαφήμιση θα μπορέσουμε νομίζω να προχωρήσουμε σχετικά γρήγορα σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Λοιπόν για το roaming. Νομίζω ότι στόχος μας είναι, ο ιδανικός στόχος είναι η κατάργηση των επιβαρύνσεων οποιασδήποτε μορφής επιβαρύνσεων. Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε σχετικά καλά στο Συμβούλιο. Δεν είμαστε μόνο οι εμείς που περιμένουμε να υπάρξουν και νέοι κανόνες και για, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το θέμα είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, όπως είπα, για το ψηφιακό εμπόριο. Και στα πλαίσια του TTIP και στα πλαίσια της γενικότερης ασφάλειας των συναλλαγών των διαδικτυακών. Για το θέμα τώρα των γυναικών. Χαίρομαι γιατί οι γυναίκες κατανοούν τις ευκαιρίες τις οποίες παρέχει το ψηφιακό εμπόριο. Την Τσεχία φυσικά τη γνωρίζω καλύτερα. Να πω ότι και κατά τη διάρκεια της κρίσης το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν στη χώρα μου δημιουργήθηκαν από γυναίκες. Λοιπόν, κάθε κρίση μπορεί να είναι και μια ευκαιρία και πρέπει οι πολίτες ε, να εποφεληθούν. Λοιπόν, αυτά ε, για το TTIP. Είπαμε θα επιδιώξουμε τα υψηλότερα ε, δυνατά επίπεδα προστασίας. Δεν μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένη και εγώ πολιτικός είμαι και ε, δεν ξεφεύγω για να μην απαντήσω αλλά ξεφεύγω γιατί πρέπει να μελετήσω το θέμα και να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση. Σεβαστές οι βασικές αρχές της διαφάνειας των διαπραγματεύσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά η κυρία Μάλστρομ το TTIP δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και κλεισμένων των θυρών. Αυτό θα θεωρεί το ύποπτο. Όλοι γνωρίζουν τι δυσφορίες και τη δυστημία που υπάρχει για το TTIP και θα πρέπει λοιπόν μέσω της δεκτικότητας και της επικοινωνίας εγώ δεν ανήκω στην κεντρική ομάδα διαπραγματεύση, αλλά όταν συζητήσουν τα θέματα τη προστασία των καταναλωτών θα είμαι παρούσα. Για την εδαφικότητα τώρα και το, τις περιοχές ισχύω των πνευματικό, της πνευματικής ε, ιδιοκτησίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο άπτεται άμεσα της α, ε, ψηφιακής αγοράς. Αλλά τίθεται το θέμα αυτό και εκεί όπως επίσης και το θέμα ε, της προστασίας των καταναλωτών και η παράδοση δεμάτων. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Στην ερώτησή σας πάντως εγώ δεν μπορώ να απαντήσω άμεσα, δεν γνωρίζω την απάντηση. Λυπάμαι που τελειώνω ε, λέγοντας για ένα θέμα ότι δεν ε, ξέρω να σας απαντήσω. Πάντως σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σας. Ανταλλαγή απόψεων για το κείμενο, την γνωμοδότηση του Πασκάλ Μπιουγάν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πασκάλ, Μπορεί, θες να πάρεις το λόγο. Αν σε έβλεπα, ε, θα ήταν και καλύτερο. Κυρίες μου, φύγετε από τη μέση. Ευχαριστώ, Βίκη, που μου δίνεις το λόγο. Πρόκειται για μια ανταλλαγή απόψεων, έτσι το λέμε αυτό. Ε, θα προσπαθήσω να ακούσω παρά να εκφράσω την άποψή μου. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι κάναμε ανταλλαγές απόψεων με τους κοιόδης συζητητές για αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και συνολικά οι θέσεις είναι κοινέ. Θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία, νομίζω, αυτό επιθυμώ εγώ και θέλω να έχουμε και συνενετική μας συμφωνία όσο γίνεται. Δύο-τρία λόγια θα πω μόνο. Η φιλοσοφία η δική μας, κοινή φιλοσοφία είναι, είναι ότι υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις αυτές δεν θα πρέπει να γίνουν όπως να είναι και όπου να είναι. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα κονδύλια του ορίζοντα 2020 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα πρέπει να σέβεται τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ισχύον και εκτιμένο. Αυτό το λέμε όλοι. Στα πλαίσια του άρθρου 1.1. Εγώ θέλω να αναφέρω τις μικροεπιχειρήσεις, τις ε, κοινωνικές επιχειρήσεις και τις ε, επιχειρήσεις αλληλεγγύης για να διευρύνουμε λιγάκι το πεδίο του άρθρου. Θέλουμε να υπάρχει μια προστέμενη κοινωνικο-οικονομική και περιβαλλοντική αξία και μακροπρόθεσμα και θέλουμε ε, να μιλήσουμε εδώ για τις επιχειρήσεις που έχουν λιγότερους από 1.500 ε, εργαζομένους. Αρχικά ήταν 1.000 εργαζόμενοι. Γιατί πήγαμε στους 1.500. Δεν θέλω να υπάρχει αμφισημία εδώ. Δεν είναι ότι επειδή μιλάμε για 1.500 ε, εργαζόμενους, οι υπόλοιπε επιχειρήσεις δεν μπορούν να κάνουν αιτήσει. Όχι. Ε, υπάρχει και το 5 5.2. Στα πλαίσια αυτού μπορούν να... 102, συγγνώμη. Οι μικρές επιχειρήσεις, 1.500 εργαζόμενοι όμω, είναι ο ορισμός που υπάρχουν στι κατευθυντήριε γραμμές της Ένωσης για τις ε, κρατικές ενισχύσεις. Με σκοπό να προωθήσουν τις ε, επενδύσεις ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το λέω αυτό για το ΕΛΚ που έκαθε το ερώτημα. Γιατί 1.500 εργαζόμενοι. Η απάντηση είναι για να σεβαστούμε τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, άρθρο 102 η ολοκλήρωση της ε, ενίας αγοράς, ψηφιακής ενίας αγοράς, ε, δημόσιες υπηρεσίες. Θα πρέπει ε, τα project αυτά να προωθούν αυτές τις επιχειρήσεις και τους βιώσιμους και τις βιώσιμες διώσιμες μεταφορές. Θα πρέπει να γίνει επίσης ε, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική μελέτη για τα project που επιλέγονται. Θα πρέπει να έχουν θετική επίπτωση στην απασχόληση και να εμπλέκουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και αυτό πολύ σημαντικό. Ε, υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι αρχές θα πρέπει να σεβαστούν όσο μπορούν τα νέα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια για την ανάθεση των ε, δημοσίων συμβάσεων. Αυτά πολύ σύντομα για να μην καθυστερούμε περαιτέρω, γιατί καθυστερήσαμε προηγουμένως, οι προθεσμίες. Αύριο έχουμε ένα νέο ραντεβού των σκιωδών στη μία η ώρα για να συζητήσουμε τους συμβιβασμούς και θα ψηφίσουμε την επόμενη Τρίτη. Όλα αυτά δηλαδή είναι επίγοντα, πιέζουν. Και ελπίζω ότι πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε τελικούς συμβιβασμούς. Ευχαριστώ. κυρία Παουνόβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Εκ μέρους ε, του κυρίου Στέφανιτς που είναι ο σκιώδης εισηγητής μας, καλωσορίζουμε την πρόταση της Κομισιόν για την πρόθεση των επιχειρήσεων και την αυξημένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις ο κύριος Στέφανης καλωσορίζει την εστίαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γιατί παίζουν ε, βασικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και είναι κυρίως αυτές που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι οι κύριοι, δικαιούχοι το, της υποστήριξης που προβλέπεται στα πλαίσια της πρότασης. Προτείνει επίσης προσθήκες στο άρθρο 5.2 για να συμπεριλάβουμε και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, κυρίως ε, της ε, ψηφιακής ενίας αγοράς και των ψηφιακών υποδομών. Το ΕΛΚΑ καλωσορίζει την αναφορά στην ανάπτυξη της ε, ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υλοποιήσουμε τους στόχους αυτού του κανονισμού και να θέσουμε τα θεμέλια για την βιομηχανική ρόμη, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και για να υπάρξει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αντιγωνιστικότητα. Ε, ενιαία ψηφιακή αγορά και ψηφιακές υποδομές. Η αναφορά είναι πολύ σημαντική γιατί αν έχουμε τέτοια ενιαία ψηφιακή αγορά μπορούμε να έχουμε πλέον ανάπτυξη, καινοτομία, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, κυρίως για τους νέους οι ψηφιακές υποδομές για τους νέους είναι πάρα πολύ σημαντικές, είναι τεχνική προϋπόθεση. Και για τη γνώση και για μια κοινωνία που δεν αφήνει κανέναν έξω. Παράλληλα, είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση σε τομείς της ψηφιακής αγοράς που έχουν μεγάλο δυναμικό για ανάπτυξη και απασχόληση. Καλό θα ήταν όμως να αφήσουμε και κάποια ευελιξία ούτω ώστε βιώσιμα έργα σε άλλους τομείς να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο βαθμό που ευθυγραμμίζονται και σέβονται τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι να απόψή μου είναι σημαντικό να υπάρχει προσθετικότητα με άλλα μέσα και να έχουμε θετική επίπτωση των επενδύσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην υποσκάψουμε τους στόχους της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η έλλειψη ανάπτυξη των ε, χρηματαγορών σε ορισμένα κράτη-μέλη παρεμποδίζει την υλοποίηση των ε, γενικών στόχων του καονισμού. Γι' αυτό είναι σημαντικό υψηλής ποιότητας τεχνική αρρωγή να δοθεί και μέσω της αποκέντρωσης ενός συμβουλευτικού κέντρου. Ενός αποκεντρωμένου, συμβουλευτικού χώρου, πούμε. Οι τροπολογίες που θέλουν να ενισχύσουν την εσωτερική αγορά είναι πρόσδεκτες ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την ανταγωνιστικότητα, για την καινοτομία και κάποιες άλλες ε, καλές προτάσεις έχουν γίνει από άλλες ομάδες, θα τις υποστηρίξουμε και αυτές. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τροπολογίες που περιπλέκουν την ε, διαδικασία λήψης των αποφάσεων ή που πολιτικοποιούν την διαδικασία λήψη αποφάσεων προς τροπολογίες 58 και 27. Θέλουμε, υποστηρίζουμε την διαγραφή του άρθρου 18 και 19 και αν δεν υπάρχει σαφή ένδειξη για τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, θέλουμε να μην ξεχνάμε ότι οι επενδυτές χρειάζονται προβλεψιμότητα, αλλιώς δεν θα υλοποιήσουμε τους στόχους αυτού του επενδυτικού σχεδίου για την κινητοποίηση δηλαδή και ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά μας σημεία. Σημεία δηλαδή που ήθελε κυρίως ο Σκιώδης συζητητής και που σας τα διαμηνύω εγώ. Ο Σέρτζο Κονφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον, κύριο Ντάντι, ο οποίος είναι σε ταξίδι. Πάει στον Παναμά. Δεν ξέρω αν στον Παναμά έχουν και εκεί προβλήματα οι καταναλωτές. Θα μας πει όταν γυρίσει. Τέλος πάντων, εγώ πρέπει να σας πω τώρα ότι ο προσανατολισμός των σοσιαλιστών είναι σημαντικός. Εμείς θέλαμε να αυτό το έκτακτο σχέδιο επενδύσεων, γιατί το μέλλον της Ευρώπης θα είναι ένα μέλλον θετικό μόνο αν η οικονομία των επιμέρους κρατών μελών της Ένωσης επιστρέψει στην ανάπτυξη. Κάτι που δεν συνέβη τα τελευταία χρόνια. Μια μακρά περίοδο. Επομένως πρέπει να έχουμε και πόρους και να εντοπίσουμε το, το πού θα γίνουν οι επενδύσεις και το ρόλο που θα παίξουν αυτές οι επενδύσεις. Γι' αυτό θα πρέπει το Ταμείο να γίνει πάρα αυτά λειτουργικό. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και σε ορισμένες περιοχές η επιδείνωση είναι εντυπωσιακή. Η ποιότητα ζωής εκατομμυρία ανθρώπων ε, είναι σε άσχημη κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν γρήγορα και πρέπει να είναι πολύ ευέλικτη η λειτουργία του Ταμείου, ούτω ώστε να μην είναι ο όμοιρος της γραφειοκρατίας και να μην καθυστερεί και η χρήση και οι θετικές επιπτώσεις από τη χρήση του Ταμείου. Στο μεταξύ χρειαζόμαστε να εξετάσουμε με προσοχή τις περιοχές που είναι οι πιο έκθετες, που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, που είναι πολύ εύκολο να τις δούμε, έτσι, και που πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι προτεραιότητα. Προσοχή. Μην θεωρήσουμε ότι όλη η Ευρώπη είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Ακόμα και και να το κοιτάξουμε, θα δούμε ότι υπάρχουν διαφορέ. Και επίση πρέπει να δούμε ποιοι τομεί έχουν τη μεγαλύτερη δυναμικότητα, το μεγαλύτερο δυναμικό. Ε, Κυρίω οι τομεί που έχουν το, τη μεγαλύτερη καινοτομία. Αν τις ε, τονώσουμε αυτές, αυτούς τους τομείς, θα έχουμε και άμεσες ε, επιπτώσεις στην απασχόληση και στη δημιουργία πλούτου, αλλά θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε την καινοτομία αυτή, ούτως ώστε το παραγωγικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει παγκοσμίως ανταγωνιστικό. Αυτό για μας είναι το κλειδί της συζήτησης που κάναμε με τον εισηγητή, του οποίου τη δουλειά με εκτιμώ. Στη συνεδρίαση των σκιωδών τις επόμενες ημέρες θα επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα, θα ζητήσουμε το θέμα του, θα το θέμα του κατοφλίου, να το δούμε περισσότερο. 3.000 ε, εργαζόμενους ε, αναεπιχείρηση που θα πρέπει να κατέχουν σε 1.500. Εμείς δεν έχουμε ιδεολογικές προκαταλήψεις. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δούμε ποιο είναι το κατάλληλο νούμερο, γιατί η προτεραιότητα στο παραγωγικό σύστημα και των αγαθών και των ε, υπηρεσιών είναι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τα 1.500 και τα 3.000 εργαζόμενοι. Μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις και αυτά τα, αυτά τα κατόφλια μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε ό,τι αφορά το παραγωγικό ιστό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να διαλέξουμε ένα κατόφλι ε, λαμβάνοντα υπόψη όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές, ούτως ώστε να μην αποκλείσουμε επίτηδες καμία περιοχή ή να μην μειώσουμε την παρέμβαση στη συγκεκριμένη περιοχή έτσι αθέλητα. Μόνο και μόνο επειδή δεν μετρήσαμε σωστά τις ε, διαστάσεις στη συγκεκριμένη χώρα ή στη συγκεκριμένη περιοχή και τα νούμερα τα οποία έχουν νόημα. Επίτα, κάποια θέματα που ενδιαφέρουν πολύ τους ε, σοσιαλιστές. Το σωστό εντοπισμό των τομέων που έχουν το μεγαλύτερο καινοτόμο δυναμικό, που μπορούν να δημιουργήσουν δηλαδή, και να διαδώσουν θετικές, επιπτώ, ε, θετικές επιπτώσεις ε, που παράγονται από τα κέρδη. Και να δώσουμε μεγάλη προσοχή στη σχέση ιδιωτικού δημοσίου τομέα οι δημόσιες επενδύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές όπως είναι η φιλοσοφία του, σχεδίου αν παρασύρει ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Οι προβλέψεις, οι εκτιμήσεις που κάνει η Κομισιόν νομίζω έχει, έχει υπερβολές. Το να δημιουργήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις, αυτά που λέει η Κομισιόν μου φαίνονται λίγο αξιόπιστα. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε δημόσιους τομείς που είναι σε θέση να κάνουν τη διαφορά και να παρασύρουν τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις, ούτως ώστε το συνολικό αποτέλεσμα να είναι όσο το πιο καλό. Ευχαριστώ εκ νέου τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε, για τη διαθεσιμότητά του και επαναλαμβάνω, έχουμε την πρόθεση να συνεργαστούμε, ούτω ώστε να φτάσουμε πολύ γρήγορα, εμπρόθεσμα, σε μία λύση, η οποία να είναι η πιο πλήρης και να την συμμεριζόμαστε όλοι μας. Ευχαριστώ. Um, Σας ευχαριστώ. Είμαι σκιώδης από την ομάδα του, του e ECR. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή που εξασφάλισε ότι είναι πραγματικά εστιασμένη η έκθεση. Και ότι διασφάλισε ότι θα μπορούσε να ακουστεί και η φωνή της ΣΥΜΚΟ στο θέμα αυτό. Ήταν πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Είναι προφανές ότι η Επιτροπή Μεταφορών θα είχε άποψη όταν αναφέρεται ρητά το θέμα των μεταφορών ή ότι η Επιτροπή Πολιτισμού, η Επιτροπή Βιομηχανίας ήταν σίγουρο ότι θα ακούγονταν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και της Προστασίας των Γονατών σε κάποιες περιπτώσεις ε, αλληλεπικαλύπτονται. Οι αρμοδιότητες που προβλέθηκαν ήταν συγκεκριμένα για το άρθρο 5.2. Και στο άρθρο 1 το θέμα της φιλοδοξίας του ίδιου του Ταμείου. Στο άρθρο 1. Αν αρχίσουμε και συζητάμε άλλα άρθρα όπου δεν έχουμε αρμοδιότητα, Ανησυχώ ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός τροπολογιών που κατατέθηκαν με καλή πρόθεση ασφαλώς. Αυτό όμως μπορεί να υπονομεύσει την ε, τοποθέτησή μας στο σύνολό τη. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή για το γεγονός ότι στην πρώτη του τροπολογία ε, διευκρινίζει με σαφήνεια ότι θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενιαία αγορά. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν στρεβλώσεις. Μας απασχολεί πάρα πολύ η ισότητα. Γι' αυτό και έχουμε σαφεί κανόνες για τον ανταγωνισμό. Γι' αυτό όλοι είναι πολύ σαφώς ορισμένες και εξαιρέσει. Χαιρόμαστε που το διευκρινίζετε λοιπόν αυτό. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οποιοδήποτε κονδύλιο θα δαπανηθεί με μη διακριτικό τρόπο. Επίσης, το ότι εξετάζουμε από πού μπορεί να έρχονται άλλα κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό προκειμένου να συγκρίνουμε παρόμοια μεγέθη. Για να μην συγκρίνουμε, για παράδειγμα, με επενδύσεις που δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν από τον δυτικό κλάδο. Να μην συγκρίνονται αυτά με άλλους τομείς όπου οι επενδύσεις θα μπορούσαν να γίνουν από τον δυτικό κλάδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τις σχετικές τροπολογίες. Να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για μια προσωρινή λύση σαφώς, αλλά είναι μια προσωρινή λύση η οποία λειτουργεί γιατί εννοείται ως ένα ταμείο στρατηγικών επενδύσεων για να δώσει ένα έναυσμα στις επενδύσεις στην Ευρώπη οι οποίες τόσο έχουν πληχθεί από την τρέχουσα κρίση και γι' αυτό λοιπόν ως ομάδα θέλουμε να διασφαλίσουμε ως ECR ότι αυτό δεν υπονομεύει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να συνοδεύεται και από άλλες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, ιδιαίτερως από τον ιδιωτικό κλάδο και σε διαφορά τα δημόσια οικονομικά, προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη. Είναι σημαντικό λοιπόν το Ταμείο να περιλαμβάνει μια επιλογή προγραμμάτων γιατί οποιαδήποτε πολιτική διάσταση μπορεί να διώξει αυτούς τους επενδυτές που προσπαθούμε να προσελκύσουμε στη τελική ανάλυση. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε καταθέσει τραπολογίες για την επιλογή των έργων βάσει της ε, βιωσιμότητάς τους, βάσει της αξίας τους πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δοθεί εμπιστοσύνη στους ε, επενδυτές. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει αυτή η εμπιστοσύνη θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι αξιόπιστη η επένδυση. Και κάποιες από τις τροπολογίες υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένες οι, τα κονδύλια από τις ε, Ευρωπαϊκής αυτό νομίζω υπονομεύει την αξιοπιστία όλου του εργαλείου και δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει τη λύση. Αν θέλουμε να λειτουργήσει το ΕΦΣΥ, θα πρέπει να φροντίσουμε να γνωρίζουμε ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου. Αν υπάρχει ανάγκη να προέλθουν χρήματα και κονδύλια από τον προπολογισμό για την έρευνα, να μην προέλθει από τους βασικούς τομείς, να προέλθει από τομείς όπου υπάρχει ήδη, για παράδειγμα, σύμπραξη δημοσίου τομέα. Προφανώς θέλουμε να δούμε πιο πολλά, πιο πολλές επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στις υποδομές, στην ψηφιακή ενιαία αγορά, στις σχετικές υποδομές και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της μόχλευσης, ε, ελπίζουμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για το έργο σας. Γι' αυτό λοιπόν ε, συνεχίστε παρακαλώ να μας ενθαρρύνετε προκειμένου να παραμείνουμε εξίσου εστιασμένοι γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάποιες τροπολογίε ενδεχομένω να αποδυναμώσουν το μήνυμα που θέλουμε να αποστείλουμε ω Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ τον εισηγητή μας. Πρέπει να βελτιωθεί το επενδυτικό περιβάλλον. Απαιτείται όμω για να γίνει κάτι τέτοιο νοπό κεφάλαιο. Και αυτό είναι το κλειδί. Δεν βλέπω τα χρήματα πουθενά Μιλάμε για υψηλά επίπεδα μόχλευσης, καλό θα ήταν, αλλά οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν θα έλθουν μόνο και μόνο λόγω της υψηλής μόχλευσης. Θέλουν να δούνε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε χώρες που έχουν αναλάβει υποχρεώσεις και είναι έτοιμες να μεταρρυθμίσουν. Υπάρχουν πολλές τέτοιες χώρες οι οποίες ακολουθούν την πορεία αυτή. Δεν έχει νόημα ε, το να κυνηγάει κανείς το χρήμα όταν το χρήμα δεν θέλει να έρθει. Πρέπει να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη τα οποία είναι προοδευτικά, τα οποία προχωρούν και όσο πιο ευφυείς είμαστε στην εφαρμογή των διαφορετικών αλλαγών τόσο περισσότερα θα είναι ε, τα διαθέσιμα. Νομίζω ότι είναι μια αφορμή για τις χώρες ε, για να μπορέσουν να μεταρρυθμίσουν ε, με μεγαλύτερη προθυμία. Είχαμε αποφασίσει την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά και με τις δικές μας αρμοδιότητες. Εγώ έχω κάνει τροπολογίες στα άρθρα 1 και 5 Έχω συγκεκριμένες απόψεις όμως και για την διακυβέρνηση του συγκεκριμένου αυτού ταμείου. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Έχει σημασία επίσης να δούμε με ποιο τρόπο θα εργαστούν όλα αυτά. Αν πετύχουμε τον στόχο με τη μόχλευση, απαιτείται μια πολύ ισχυρή επιτροπή απαιτείται ακριβώς να υπάρξει μια σωστή διαδικασία για να μπορέσει να εργαστεί το ταμείο αυτό. Οι τροπολογίες μου στο άρθρο 1 έχουν σαν στόχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σαν συνομοθέτες να αξιολογήσουν την συμφωνία που υπέγραψε η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά τα προγράμματα. Τα προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να είναι υψηλού κινδύνου. Αυτό είναι το βασικό εδώ. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν όπως είπα ευφυείς σε σχέση με το τι εννοούμε. Υψηλού κινδύνου σημαίνει υψηλές αποδόσεις. Όταν μιλάμε λοιπόν για τέτοιου είδους ε, ε, αποδόσεις, μιλάμε για αποδόσεις πάνω, για επενδύσεις υψηλού κινδύνου, μιλάμε για αποδόσεις άνω του 10%. Και τα ιδιωτικά κεφάλαια θα θέλουν τέτοιου είδους υψηλού επίπεδου αποδόσεις. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει συγχρονισμός των ενεργειακών συστημάτων. Η αγορά της ενέργειας είναι βασική μας προτεραιότητα και θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε εδώ έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη όθηση, να υπάρξουν μεγαλύτερες ε, δυνατότητες θα βοηθήσει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ε, και θα βελτιωθεί η αποδοτικότητα της ενέργειας αν μπορέσουμε να την συντονίσουμε. Νομίζω ότι αυτές είναι μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας που θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Δεν έχω άλλες παρατηρήσεις στην παρούσα φάση. Είμαι στη διάθεση των εισηγητών και των σκιωδών αύριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων για αυτά που μόλις είπατε. Για το ότι μας κατευθύνεται. μας πιέζετε να είμαστε πιο εστιασμένοι. Εγώ το κάνω μέσω των τροπολογιών μου. Δεν θέλω να προκαλέσω και να κάνουμε μια ενδελεχή συζήτηση για το αν είναι κατα καλό αυτό το εργαλείο. Είναι περίεργο που η, η Κομισιόν λέει ότι δεν μπορούν να το κάνουν λόγω της λιτότητας. Ενώ αν συνεισφέρουν και βάρουν λεφτά σε ένα ταμείο, λες και εξαφανίζονται οι νόμοι της ε, λιτότητας. Ε, δεν μπορούν να κάνουν επενδύσεις, ας πούμε, λόγω των σφιχτών προϋπολογισμών. εγώ δεν το, δεν το αναφέρω. Αυτό το αφήνω παράμερα. Δεύτερο, μόλις λάβαμε μια κρίσιμη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε τώρα με δημόσια κονδύλια ρίσκο ιδιωτικό που τα κέρδη θα μπουν στις τσέπες των ιδιωτών, ενώ εάν υπάρξουν ε, απώλειες εδώ κονδυλίων, θα χαθούν δημόσια κονδύλια. Δεν έχω υποβάλει σχετικές τροπολογίες, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό εδώ, το οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε στην νομοδότηση. Αυτό που προσπάθησα να απαντήσω, να θίξω, είναι δύο πράγματα και μία παρατήρηση. Καταρχάς, με μεγάλη χαρά άκουσα την προσέγγιση του ΕΛΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήταν και μία από τις δικές μου τροπολογίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι η πρώτη, ο πρώτος και κύριος ε, δικαιούχος αυτού του επενδυτικού σχεδίου και ελπίζω να το πούμε αυτό. Έχουμε κάνει πολλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ στην Επιτροπή μας και είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Το δεύτερο είναι το θέμα της διαφάνειας. Το ανέφεραν και οι φιλελεύθεροι όταν μίλησαν για τη διακυβέρνηση. Αλλά και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να δώσουμε σημασία στη διαφάνεια. Είναι σημαντικό, ε, είναι προς το συμφέρον μας να μην έχουμε έργα τα οποία είναι προβληματικά. Θέλουμε να ελέγχουμε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα θέμα την Τράπεζα Επενδύσεων. Και η ΕΚΟΝ θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα και πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα της ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Τελευταίο, τελευταίο θέμα η παρατήρηση. Ανησυχούσα για το ότι από τα μία καινοτομία θα πρέπει να αντλήσουμε κονδύλια. Είναι πολύ σημαντική η καινοτομία και το Ταμείο Καινοτομία και για την εσωτερική αγορά. Και Βίκη, συμφωνώ με αυτό που είπε, ότι πρέπει να υπάρξει ένα πάντρεμα κάπως, ένα συντέριασμα, γιατί αλλιώς ε, εάν δεν ε, συμμετάσχει και το ε, Ταμείο αυτό καινοτομία, κάπου θα χάσουμε. Κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει, κυρία Κάλλας. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω αυτά που είπε ο συνάδελφο. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, αν ε, υιοθετηθεί η σωστή νομοθεσία, μπορεί να προσελκύσει οι ιδιωτικές επενδύσεις. Υπάρχουν πολλά έργα που έχουν μακροπρόθεσμους κινδύνους και αγωνίζονται να προσελκύσουν χρηματοδότηση, αλλά ε, λόγω των οικονομικών δυσκολιών υπάρχουν προβλήματα. Παραδείγματο χάρη τα ευρυζωνικά έργα είναι ένα καλό παράδειγμα. Η εστίαση του Ταμείου θα πρέπει να αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις, αν θες να αυξήσεις την μόχλευση της χρηματοδότησης. Και όπως είπε και ο Άντων για την ε, Διευθύνουσα Επιτροπή, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι σωστοί κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων, τη διαφάνεια και την λογοδοσία της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων της, του Διοικητικού Συμβουλίου και της της Επιτροπής είναι πολύ σημαντικό για να έχουν εμπιστοσύνη οι επενδυτές. Τελευταίο και σημαντικό, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι, υπάρχουν, ότι υπάρχει χρηματοδότηση για τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Να έχουμε δηλαδή την απαραίτητη χρηματοδότηση που χρειαζόμαστε, καθώς περνάει από διάφορες φάσεις μια εταιρεία. Ε, θα πρέπει να προωθήσουμε και μια αλλαγή της νοτροπίας. Ε, τι σημαίνει επιτυχία. Πώς ε, αγκαλιάζουμε μια κουλτούρα, ας πούμε, που δέχεται τον κίνδυνο. Πρέπει να επιτρέψουμε στον κόσμο να αποτυγχάνει, να πρέπει να το δούμε αυτό, τη δυνατότητα αποτυχίας και νέας προσπάθειας. Είναι σημαντικό και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το θέμα. Η Κομισιόν άκουσε με προσοχή. Θέλει να παρέμβει. Ένα λεφτάκι και μετά θα δώσω ξανά το λόγο στον εισηγητή. Yes, thank you, madam. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευτυχώς πολλά από τα σημεία που ήθελα να θίξω έχουν ήδη α, από τις ομάδες να ευχαριστήσω τον εισηγητή που το έπραξε αυτό παρά το γεγονός ότι ακούσαμε ασφαλώς με προσοχή και διακρίναμε διαφορά στις απόψεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Τα θέματα που μας απασχολούν ιδιαίτερα, ωστόσο, να σας εξηγήσω γιατί πιστεύουμε ότι είναι τόσο σημαντικά. Καταρχάς, ασφαλώς είμαστε ιδιαίτερα που υπάρχει η αίσθηση του κατεπήγοντος, όπως είπε και ο εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Είναι κοινός τόπος πλέον αυτό. Όλοι συμφωνούμε με την ανάλυση ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επενδύσεις σε θέσεις εργασίας, επίσης ε, στην ε, Ευρώπη, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γρήγορα και ότι θα πρέπει να κάνουμε και κάτι ε, που να έχει νόημα σε ό,τι αφορά τον όγκο Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αυτή η νομοθετική πρόταση για την ε, επενδυτική πρωτοβουλία έχει ως κύριο μέλημα να δημιουργηθούν 315 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια νέες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια και να δημιουργηθούν και τέσσερις εργασίες Και αυτό να γίνει το σύντομο δυνατόν. και αν το πράξουμε αυτό, θα υπάρξει αποτυχία, θα θεωρηθεί αυτό αποτυχία από πλευρά μα. Γι' αυτό λοιπόν. Θεωρούμε ότι οτιδήποτε είναι υπερβολικά χρονοβόρο ως νομοθετική διαδικασία, αλλά και ως ε, εφαρμογή των συστημάτων που έχουμε αποφασίσει, θα πρέπει να αποφευθεί. Έχουμε προτείνει λοιπόν μια πολύ εναρμονισμένη διαδικασία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να είναι σαφές. Ναι, να συνοψίσω λοιπόν αφού δεν έχω χρόνο. Να είμαστε γρήγοροι αλλά και ευέλικτοι στη διαδικασία προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη αξιοποίηση του δυτικού κεφαλαίου. Αυτό μας απασχολεί στην εφαρμογή της οδηγίας. Και επειδή πρόκειται για δημόσια κονδύλια, ασφαλώς υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμοστούν, κάποια κριτήρια για ό,τι αφορά τι ευ... ευρωπαϊκέ πολιτικέ, σε ό,τι αφορά τη συμπληρωματικότητα, γιατί δεν έχει νόημα να δαπανηθούν χρήματα σε τομείς όπου θα υπήρχε έτσι και μια επένδυση. Είναι σημαντικό επίση να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Μία σύντομη παρα τήρηση για τις τροπολογίες που αφορούν το από πού θα προέλθουν τα κονδύλια. Καταλαβαίνουμε τη λογική αυτή. Απόλυτα. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που απέχουν περισσότερο από την αγορά και βλέποντας τις προτάσεις βλέπουμε ότι αυτό όντως γίνεται τα προγράμματα υπό τον ορίζοντα 2020 που έχουν μεγαλύτερη απόσταση από την αγορά. Διαπιστώνουμε ότι αποτελούν ποσοστό 1,7% σε σχέση με άλλα έργα τα οποία έχουν απόδοση 10% για επανατοποθέτηση στην αγορά. Ήθελα λοιπόν να το διευκρινίσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Θα συνεψίσετε. Κλείνοντας, να εκφράσω την ικανοποίησή μου που κάνω αυτή την έκθεση σε αυτήν την Επιτροπή και όχι σε άλλες. Να πω επίσης ότι είναι θετικό το ότι αποφασίσαμε να στοχεύσουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στην Επιτροπή μας ε, την δουλειά την οποία κάνουμε. Όταν άκουσα τον κύριο De να θέτει το θέμα της φύσης των επενδύσεων και των προγραμμάτων λιτότητας, Προφανώς το θέμα θα μας απασχολούσε πολύ καιρό. Λοιπόν, είναι θετικό το ότι είναι υψηλής ποιότητας η προσπάθεια η οποία γίνεται και συμμεριζόμαστε την προσπάθειά μας, στα πλαίσια της προσπάθειάς μας, μια φροντίδα να κρατήσουμε ακέραιη την αγορά, να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και να μειώσουμε και τον αριθμό των 27 εκατομμυρίων ανέργων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας τους βοηθήσουμε λοιπόν μέσα από αυτή την έκθεση αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλα για αυτό το τμήμα της συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που αντικατέστησαν άλλους συναδέλφους. Η επόμενη συνάντησή μας θα γίνει την επόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Στις 24 του μηνός, 3 το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Περνάμε αμέσως στις συνεδρίες των συντονιστών.